ντροπέ αποφάσισαν να ξεκινήσουν διαθεσμικέ διαπραγματεύσει βάσει του άρθρου 78 του ιστορικού κανονισμού. Ε, οι εντολέ για τι διαπραγματεύσει αυτέ βρίσκονται στον ιστότοπο τη Ολομέλεια και θα εκδοθούν και στα πρακτικά τη Συνόδου βάσει του άρθρου 231.4 δεύτερο εδάφιο ε,